Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση, τα πρακτικά της χθεσινής ε, συνεδρίασης και τα κείμενα τα οποία έχουν εγκεκριθεί, έχουν δημοσιευθεί, υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά. Εάν όχι, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Έχουμε πάρει τη θέση του Συμβουλίου για, σε πρώτη ανάγνωση και τη θέση της Κομισιόν. Τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του Κοινοβουλίου και υπάρχει από τη στιγμή δημοσίευσης μια προθεσμία τριών ε, μηνών για αντίρρηση σε σχέτη. Ερχόμαστε τώρα σε θέματα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου και δημοκρατίας και ξεκινάμε... Ξεκινάμε με τη βία κατά των γυναικών στην Ινδία. Καταρχήν, οι συντάκτες του ψηφίσματος. Ξεκινάμε με την κυρία Ντέλη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που η Ινδία αποτελεί αντικείμενο μια δεύτερη συζήτηση μέσα σε δύο μήνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου και παρόλα αυτά η κατάσταση των γυναικών είναι καταστροφική η σεξουαλική βία είναι πλέον κοινότυπη και έχουμε ένα βιασμό κάθε 20